ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες για την εκλογή των κοσμητόρων. Συγχαίρω όλους που εξελέγησαν. Έχουμε μία ψηφοφορία τώρα για την αριθμητική σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Έχουμε την πρόταση της διάσκεψης των Προέδρων ως πρόταση. Όσοι είναι υπέρ να σηκώσουν το χέρι τους παρακαλώ αυτής της απόφασης. Υπέρ κατά αποχές Νομίζω ομόφωνα σχεδόν εγκρίθηκε η πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Διακόπτεται η συνεδρίασή μας στην Ολομέλεια μέχρι τις 3. Ευχαριστώ.